να υπάρχει ένα πάνελ ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα παρακολουθούν την ποιότητα σε ό,τι αφορά την υλοποίηση, την εφαρμογή του κράτους δικαίου και των ε, ε, άλλων αξιών, θεμελιωδών αξιών. 158 τροπολογία θα μας έκανε να επαναχωρήσουμε και υπάρχει και 88 τροπολογία αντίστοιχη. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να βρούμε συμβιβασμό πάνω στα όσα έχουμε ήδη πετύχει μέχρι τώρα. Α, πώς να σας πω, γκαρδιαθάμπαλ, το ρουμπιάλ μου φαίνεται πιο εύκολο, τέλος πάντων το πάρεις προσωπικά. Αυτό απέλεξε λοιπόν είναι τι γίνεται αν ε, ο μηχανισμός ενεργοποιείται. Και φτάνουμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Για παράδειγμα, στην Ουγγαρία, το Φίντες, στον τη διαχείριση των κονδυλίων, χρησιμοποιεί αυτό και ως μέσο άσκηση πολιτικής επιρροής ε, για τη δημιουργία πολιτικής ισχύω. Θα μπορούσε να υπάρχει δυνατότητα σε έτσι περίπτωση αρκετά ακραία, να υπάρξει μεταφορά των κονδυλίων στην Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή. Δηλαδή, αν ενεργοποιηθεί ο μηχανισμό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να κινητοποιηθεί η μηχανή των τοπικών αρχών, τοπικών ΜΚΟ κατά της Ένωσης, που λένε ότι με αυτό το εργαλείο τους ε, στραγγίζουμε, στεγνώνουν από κοινοτικά κονδύλια. Δηλαδή, δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε τις τοπικές αρχές ή επιχειρήσεις ή ΜΚΟ που έχουν καλέ πρωτοβουλίε. Θέλουμε τη διαχείριση των κονδύλων να την αφαιρέσουμε από την κυβέρνηση ε, που δεν σέβεται τι θεμελιώδει αξίε. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η δυνατότητα προκειμένου να αποφευχθεί ότι με την επιβολή των θεμελιωδών αραρχών όπω είναι το κράτο δικαίου να δημιουργούμε ένα ισχυρό όπλο ε, που στρέφεται κατά αυτών που δημιουργούν στην Ευρώπη και τους οποίους τους στερούμε από χρηματοδότηση. φορολογία τώρα, κατά πόσο πρέπει να ενταχθεί σε όλο αυτό το τη συζήτηση και το διάλογο για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Είχαμε το σκάνδαλο Κουμέξ με τα μερίσματα και κάποια από τα μέτρα τα φορολογικά βλέπουμε ότι είναι βαθιά ριζωμένα στην κακοδιαχείριση και στην έλλειψη του κράτους δικαίου. Άρα νομίζω ότι είναι απόλυτο σκόπιμο να το συμπεριλάβουμε το θέμα της φορολογίας. Σας ευχαριστώ για το έργο σας και περιμένω και την ε, συνάντηση μεταξύ των σχεδόν εισηγητών όπου μπορούμε, πιστεύω, να σημειώσουμε περαιτέρω πρόοδο. Κύριε Αλή. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι αγαπητοί εισηγητές. Η αναγκαιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να παράγει το απαραίτητο έργο με βάση προτεραιότητέ, τη έχει κρίσιμη σημασία την σύγχρονη εποχή, δεδομένου ότι περνάμε στο νεο πολιτισμικο δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027. Όπω υπογραμμίστηκε ήδη, όλες αυτές οι προποθέσει έχουν να κάνουν με την τήρηση των αρχών του κράτου δικαίου. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να σημειώσω ότι καλωσορίζουμε την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεδομένου ότι το κείμενο αυτό παρουσιάζει ένα νομοθετικό πλαίσιο επιτυχία για το... την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ιδιαίτερα υπογραμμίζει το πόσο σημαντική είναι η τήρηση και εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού σε κάθε στάδιο τη λειτουργία του και λαμβάνομενων υπόψη των τροπολογιών που προτείνονται με το κείμενο. Υποστηρίζουμε ιδιαίτερα την έμφαση που δίδεται στην ε, τήρηση του κράτους δικαίου και των θεμελιδών δικαιωμάτων και τα συναφή, τους συναφείς ορισμούς ιδιαίτερα θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικές ε, οι διατάξει που αναφέρονται στα μέτρα αυτά, ιδιαίτερα όσον αφορά το κράτο δικαίου και κράτο ε, μέλο που μπορεί να επηρεάζει τι αρχέ τη ε, χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ανάγκη και δημιουργία πρώτον ενό μηχανισμού που θα είναι το δυνατόν πιο σαφής ευθυγραμμισμένος αλλά και θα εξασφαλίζει την προστασία των ε, δικαιούχων και ταυτόχρονα υπάρχει ανάγκη για έναν επικοδομητικό διάλογο που θα πρέπει να οργανώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίσης <laughs> πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάγκη να ε, παρακολουθούνται εκ του σύνεγγες οι κατευθυντήρες Ο κανονισμό θα πρέπει να είναι σωματωμένος στο νέο πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο και βεβαίω θα συνεχίσουμε και εμεί με τις επικοδομητικές μας προσπάθειες. Σα ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Στά είναι ο είναι αλλά νομίζω το έχει καλύψει ο κύριος Γκίγκολτ που τα είπε όλα. Καλώ ευχαριστώ. Λυπή. Κύριε Ντόιτς. Ε, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, για να συντομεύω θα ήθελα να συντομέψω τα καλωσορίσματα και τις ευχαριστίες για ένα θέμα όμως πάρα πολύ σημαντικό που έχει να κάνει με την ποιότητα του έργου των εισηγητών. Αγαπητοί συνάδελφοι, επί της ουσίας η πρόταση αυτή εγκαθιδρύει μια διαδικασία μη ισορροπημένη. Μια διαδικασία που αντιπαρέρχεται το άρθρο 7, πράγμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και επίσης ε, στηρίζεται σε μια παρεξήγηση που λέει ότι οι στερήσεις ως προς την τήρηση των αρχών του κράτους δικαίου μπορούν να εξετάζονται σε επίπεδο του ίδιου του κράτους μέλους. ή μόνο συγκριτικά, με μια μελέτη συγκριτική μεταξύ της κατάστασης στα κρατη Όλη αυτή η διαδικασία δεν έχει καμία νομική βάση δε. Και όλα αυτά δεν είναι προσωπική μου γνώμη. Όλα αυτά που σας ανέφερα, τα τέσσερα σημεία, είναι η γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου για την πρόταση της Επιτροπής. Τα ξαναλέω. Νομική υπηρεσία του Συμβουλίου θεωρεί ότι δεν είναι ισορροπημένη η πρόταση, θεωρεί ότι αντιπαρέρχεται το άρθρο 7, άρα έχει νομικό ελάττωμα και δεν έχει επαρκή ούτε τεχνική ούτε και νομική βάση. Φρονώ δε ότι παρά είναι... Θα ήταν μεγάλη πολυτέλεια να αναμιλάβουμε υπόψη αυτήν την ε, γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου. Εάν μια πρόταση δεν αντιστοιχεί σε κανόνες δικαίου, με όλες τις καλές προθέσεις που μπορεί να μπνέουν τους εισηγητές, δεν μπορεί να προχωρήσει. Και ξέρω ότι αυτή τη στιγμή εγγράφαμε στη μειονότητα μετά όσα λέω. Ξέρω ότι δεν είναι του σειρμού η πρότασή μου, αλλά ε, καθώς είμαι αγωνιστής των ανθρωπινών δικαιωμάτων εδώ και 30 χρόνια, μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητας ότι μόνο με εργαλεία του κράτους δικαίου μπορεί να προστατέψει κανείς το κράτος δικαίου. Εδώ λοιπόν η πρόταση αυτή δεν μας εξασφαλίζει ούτε το ελάχιστο επίπεδο τήρησης των αρχών του κράτους δικαίου με τις διαδικασίες που προτείνει. Και οι τροπολογίες δεν αποκαθιστούν το πρόβλημα που στη βάση του είναι πως όλη αυτή η διαδικασία έχει στηριχθεί σε προϋποθέσεις σε στοιχεία και προαπαιτούμενα η βάση που δεν μπορεί να αναγνωριστεί ως κράτος δικαίου. Για δε την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάντα τα μέτρα που θα λαμβάνονται πρέπει να είναι αναλογικά. Η αντιστροφή του βάρους της απόδειξης είναι απαράδεκτη. Ποιο θα καλείται λοιπόν να αποδείξει κάτι, γιατί τώρα έχουμε να κάνουμε με πολιτικές κατηγορίες, όχι νομικές κατηγορίες, στις οποίες καλούνται να λογοδοτήσουν τα κράτη-μέλη. Δηλαδή μιλούμε για αντιστροφή του βάρους αποδείξεως. Πρέπει να αποδειχθεί το πώς ε, ο εντοπισμός ελλείψεων ως προς το κράτος δικαίου σε ένα κράτος μέλος προκύπτει και αποδεικνύεται σε σύγκριση με το ε, με την τήρηση των αρχών του κράτους δικαίου στα λοιπά κράτη-μέλη ή σε κάποια άλλα κράτη-μέλη. Ξέρω ότι είμαι στο μειονότητα, αλλά δεν μπορώ να ε, σοπίσω και να δεχθώ αυτές τις προτάσεις. Σα ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ κύριε Σόλμπριχ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ω ε, ε, του ΠΔΠ είχαμε υποστηρίξει την ιδέα ως στοιχείο βεβαίως της δέσμης του ΠΔΠ. Είναι ένα στοιχείο μέσα στην ευρύτερη δέσμη του ΠΔΠ. Δεν είναι ανεξάρτητο μέσο, αυτό ήθελα να, να διαφημίσω. Δηλαδή κινείται εκ προς το ΠΔΠ. Και πρέπει να είμαστε σαφέστατοι σχετικά με την προετοιμασία οποιοδήποτε μέσου που θα είναι ενισχύ για τα 27 κρατη Δεν είναι κάτι που θα ισχύει προσωρινά για την Ουγγαρία ή τη Ρουμανία ή την Πολωνία. Θα ισχύει για όλους, γιατί παντού μπορεί να υπάρχει ελάττωμα της λειτουργίας του κράτους δικαίου. Τώρα βέβαια η κατάσταση διαφέρει ως προς το εξής. Έχουμε το άρθρο 7 της συνθήκη, που υποχρεώνει να αναλάβουμε κάποιο μέτρο εφόσον διακόπτεται η ομαλή λειτουργία του κράτου δικαίου. Τώρα γνωρίζουμε ότι πρόκειται για ένα μέσο που δεν προσφέρει πρακτικές λύσεις και ότι χρειάζεται ομοφωνία. Αλλά ένα μέσο θα πρέπει να είναι αποτελεσματικό και χρειάζεται άμεση αντίδραση του δικαστηρίου. Εγώ συμφωνώ λοιπόν ότι τα νομικά μέσα πρέπει να επιλύονται με νομικό τρόπο, αλλά στην πράξη αυτό δεν συμβαίνει εύκολα, ούτε αρκετά γρήγορα. Η άλλη δυνατότητα είναι να αντιδρούμε, και αυτό είναι ο το πι δελτα πι, να αντιδρούμε χρησιμοποιώντας, μάλλον, εφόσον θεωρούμε ότι οι ευρωπαϊκοί δημόσιοι πόροι, τα δημόσια κονδύλια, είναι εν κινδύνο τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Ιδάλω, θα μπορούσε κανεί τον, τον ευρωπαϊκό προπολογισμό να τον χρησιμοποιεί για οτιδήποτε. Για οποιαδήποτε παράβαση του οτιδήποτε. Και δεν είναι κατάλληλο μέσο ως ε, απόλυτη εργαλειοθήκη για οποιοδήποτε πρόβλημα. είναι πιο σημαντικό για τους δικαιούχους, μάλλον για τους αποδέκτες παρά για τους καθαρούς συνεισφορείς το θέμα. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί με τη χρήση των δημοσίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επαναλαμβάνω, να μην το χρησιμοποιούμε για οτιδήποτε, γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν θα υπήρχε και λόγος να το συσχετίσουμε με τη δέσμη του ΠΔΠ. Άρα πρέπει να ορίσουμε πάρα πολύ σαφώς το στόχο, το σκοπό του μέσου. Γιατί εάν δεν το κάνουμε δεν θα γίνει αποδεκτό από το Συμβούλιο. Γιατί αναφερθήκατε στη νομική βάση, αλλά η έλλειψη ή η ύπαρξη της νομικής βάσης για τον κίνδυνο, για τους δημόσιους πόρους και τη δαπάνη τους είναι σαφής. Άρα λοιπόν λέω πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το μέσο αλλά πρέπει να το ε, χρησιμοποιήσουμε με μια επιχειρησιακή σαφήνεια που να ρυθμίζει, να διαχειρίζεται και το χρόνο στον οποίο πρέπει να αντιδράσουμε. Γιατί αν πάμε σε ένα θέμα πολιτικού διαλόγου, πολιτική συζήτηση, κάποια τμήματα του Κοινοβουλίου θα συμφωνήσουν, κάποια άλλα θα διαφωνήσουν κτλ. Το να παρακάμπτει κανεί του κανόνε όμω, δεν είναι θέμα πολιτική τοποθέτηση. Αν τηρείς τους κανόνες του τηρείς, αν δεν τους τηρείς, δεν τους τηρείς. Και αυτό θα πρέπει να ισχύει για όλου. Αν ανοίξουμε την πόρτα σε πολιτικέ ερμηνείε και τοποθετήσει, πάει. Το θέμα χάθηκε. Γιατί θα έχουμε αέναε συζητήσει χωρί κανένα αποτέλεσμα. να χρησιμοποιείται αυτό το μέσο εφόσον υπάρχει κίνδυνος, απειλή για το δημόσιο χρήμα. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Έχουμε εδώ έναν συνάδελφο από την ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Budget, τον κύριο Βίλμπροκ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μήπως θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να μην ε, μακρηγορήσω, δεν θέλω να σας καθυστερήσω. Απλώς να πω ότι στο πάνελ των εμπειρογνωμόνων να επαναλάβω δηλαδή και την τοποθέτηση του Αντιπροέδρου Τίμερμανς όταν συζητήθηκε το θέμα αυτό. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα με τις πηγές της εμπειρογνωμοσύνης για τα ελαττώματα του Κατζικαίου σε συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό που έχουμε αντίρρηση είναι αυτό το πάνελ των εμπειρογνωμόνων γιατί θα καθιστούσε λίγο ασαφές το, το είναι τελικός αρμόδιος και υπεύθυνο. Και για τα θέματα κράτους δικαίου είναι η Κομισιόν που είναι αρμόδια για να σας αναφέρει και από εκεί πέρα εσείς να αποφασίσετε πρέπει να κάνετε. Επομένως ε, το θεσμικό, η θεσμική δομή του πράγματος αυτού πρέπει να είναι σαφής. Δεν έχουμε καμία δυσκολία να αναγνωρίσουμε από πού αντλούμε την εμπειρογνωμοσύνη για να φτάσουμε στην απόφασή μας, αλλά για αυτό που σας είπα, την δομή αυτή. Επίσης υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογή και όπως κινούνται οι συζητήσεις στο Συμβούλιο ε, πηγαίνουν προς την κατεύθυνση ότι οποιαδήποτε διεύρυνση θα ήταν προβληματική. Γιατί θα αποδυνάμωνε τη νομική βάση και θα αύξανε τις πιθανότητες επικάλυψης με το άρθρο 7. Η πρόταση ω έχει αποφεύγει αυτό το πρόβλημα επικάλυψης διότι υπάρχει διαφορετική διαδικασία από τις διαδικασίες παράβασης για παράδειγμα τύπο το άρθρο 7. Για την αναλογικότητα και το βάρος απόδειξης συμφωνούμε απολύτως η αναλογικότητα πρέπει να τηρείται πάντοτε και πράγματι πρέπει να υπάρχει το βάρος του αποδείξεως ώστε να μην υπάρχει ζημία για τον προϋπολογισμό. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για την πρόταση της Επιτροπής. Σας ήταν καλό να γυρίσουμε στους ε, δύο συνεισηγητές, Άιντα, για να ολοκληρώσουμε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν θα ανοίξουμε εδώ συζήτηση, γιατί δεν έχουμε και το χρόνο, νομίζω, αλλά δύο σχόλια ήθελα να κάνω. Καταρχάς για τον στόχο του κανονισμού. Εγώ κατανοώ τα σχόλια των συναδέλφων και τον κύριο Όλμπριχτ. Συμφωνώ δηλαδή για τον σχετισμό με το ΠΔΠ, αλλά για τη διεύθυνση ή μη του στόχου του κανονισμού. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε και πρέπει να διαβρύνουμε εφόσον, και αυτή είναι η απαραίτητη φράση, εφόσον η διεύνηση αυτή για τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκαλεί, καταλήγει σε πρόβλημα η απειλή για τον προϋπολογισμό. Και τότε οδηγούμαστε στο εξή ερώτημα. Γιατί ναι, εντάξει, για το κράτο δικαίου και τα ελαττώματα αυτά και όχι για άλλο πρόβλημα. Δηλαδή, μπορούμε να ιεραρχήσουμε τις, ε, τις αρχές και τις αξίες Τη Ευρωπαϊκής Ένωση. Συμφωνώ ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μέσο για τα πάντα, αλλά ναι για τις περιπτώσεις για τι οποίε η οποιαδήποτε παραβίαση έχει, ενέχει ζημία ή απειλή για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Δεν μιλούμε λοιπόν για οποιοδήποτε ελάττωμα και οποιαδήποτε έλλειψη τη λειτουργία του κράτου δικαίου, αλλά για το τμήμα εκείνο που επιφέρει ζημία ή απειλή για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Εγώ νομίζω ότι η πρόταση είναι απολύτως νομικά σαφής. Το Συμβούλιο έχει κάνει σχόλιο σε επιμέρους ε, πτυχές, τις οποίες δεν χρειάζεται εδώ να καθίσουμε να αξιολογήσουμε. Ω προς τα αρμοδιότητες υπό το άρθρο 7 δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η στόχευση μπορεί να είναι ίδια, αλλά η εφαρμογή μπορεί να είναι πολύ διαφορετική. Το άρθρο 7 μιλάει για τι αρμοδιότητες που πρέπει να έχουν τα κράτη-μέλη. Εδώ μιλούμε για κακοδιαχείριση των πόρων του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού υπό τις αρχές και τις αξίες τη Ευρωπαϊκής Ένωση. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αρμοδιότητα. όλα αυτά είναι πολύ σαφή. Τώρα, με τις τροπολογίες και με την τελική συμφωνία που θα υπάρξει, ίσως να περιπλακεί η συζήτηση με το Συμβούλιο, ίσως, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να μείνει στις δικές του προτεραιότητες και τα δικά του κριτήρια. Και το Συμβούλιο στα δικά του. Και αντιστοίχω θα διεξαχθεί ένα διάλογο. Δεν μου φαίνεται ευφυέ από πλευρά μα να λέμε ότι εφόσον το Συμβούλιο δεν θα δεχθεί το Α ή το Β, εμεί δεν θα τα κάνουμε. Τα οποία μάλιστα είναι και θέματα προτεραιότητα για εμά. όπως στι περιπτώσεις των ε, φορολογικών απατών, είχαμε κάνει τρεις επιτροπές στο Κοινοβούλιο για να συζητήσουμε για το θέμα. Δεν μου φαίνεται καθόλου ε, σοφό να μην θέτουμε αυτά τα προβλήματα επειδή το Συμβούλιο δεν θα τα δεχθεί. Και επαναλαμβάνω, στο μέτρο που όλα αυτά συνδέονται με τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Προεπολογισμού. Και όχι για οποιαδήποτε πρόταση έρχεται στο τραπέζι. Αυτά. Uh, Σας ευχαριστώ. Πέτρη. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω κι εγώ να ευχαριστήσω πολύ τους συναδέλφους. Με μεγάλη προσοχή άκουσα τα σχόλια. Θεωρώ ότι πια πρέπει να στιάσουμε την προσοχή μας στα ακανθόδη ζητήματα του της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής. Και επιτρέψτε μου λίγο να μιλήσω για αυτά που κανείς δεν μιλάει. Ας το σκεφτούμε λοιπόν πολύ προσεκτικά όλοι όσοι είμαστε εδώ. Εάν στη συμβαστική υπαριθμών 2 και στους ορισμούς, γιατί πρόκειται για το άρθρο 2 της πρώτας επιτροπής, προτείνουμε πρώτον το κράτος δικαίου να γίνεται αντιληπτό ως ένα άρθρο το οποίο παραπέμπει στις αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της συνθήκης αλλά και της, ε, των αρχών της Κοπενχάγης ε, διαφάνεια κράτος δικαίου, πλουραλιστικές διαδικασίες για την εγκαθίδρυση της νομοθεσίας, ασφάλεια δικαίου, παρα, ε, απαγόρευση αυθαίρετης άσκησης της εξουσίας, της Κρατική εξουσίας, ανεξαρτησία των δικαστηρίων, κρίση ανεξάρτητων θεμελιωδών δικαιωμάτων, ισότητα ενώπιον του νόμου και γενική αποτελεσματικότητα ω προς την ε, τήρηση του κράτους δικαίου που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ε, πρακτικές των, κρατών, ε, των κρατικών υπηρεσιών, των δημόσιων υπηρεσιών που μπορούν να επηρεάζουν τις αξίες της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων εκείνων που προέρχονται από μειονότητες, αξίες που είναι κοινέ στα κράτη-μέλη, στις κοινωνίες με τον πλουραλισμό, την μη διάκριση, την ε, διαλλακτικότητα, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αρχές επικρατούσες, τότε δεν μπορεί να γίνεται λόγος για κράτος δικαίου. Αυτό λοιπόν που λέω εγώ είναι ότι αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι κρίσιμα, νομίζω, είναι κρίσιμες διατάξεις. Και νομίζω ότι όντως εμείς το Κοινοβούλιο δεν πρέπει να ξεκινούμε με υποθέσεις του τι μπορεί να εγκρίνει το Συμβούλιο ή τι μπορεί να περάσει από την Επιτροπή. Τη δουλειά μας θα την κάνουμε εμεί και μόνοι μας. Αλλά ταυτόχρονα όταν κάνουμε τη δουλειά μας ως Κοινοβούλιο, εδώ μιλάμε για ένα πολύ κρίσιμο νομοθέτημα. Και πρέπει να προχωρήσει. Ξέρουμε πολύ καλά τι θέλουμε όλοι να έχουμε ολοκληρώσει πριν το 2019, πριν να αναλάβει το νέο Κοινοβούλιο, η νέα Επιτροπή κυρίως. Άρα εδώ εάν διευρυνθούν οι ορισμοί στο τομέα των αξιών αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι όχι ότι μπορεί να το τραβήξουμε λίγο περισσότερο είναι ένα άσπρο ή μαύρο δηλαδή είμαστε στο ε, όριο του, του γκρεμού και στεκόμαστε και το μαζεύουμε και ξαναχτίζουμε όλη την αυτή ή κατακρινιζόμαστε αυτό είναι το πρόβλημα που έχω εγώ ως συνεισηγητής. Νόμιζα ότι ο κύριος Γκίγκολτ μίλαγε αντί για σένα Μπάρτ σήμερα. Ευχαριστώ κύριε Evans ή κυρία Τζιλ Evans συγκεκριμένα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Από ό,τι φαίνεται Υπάρχουν ήδη κάποια σχέδια τροπολογιών συμβιβαστικών. Άκουσα να διαβάζετε κάποιο κείμενο, αν κατάλαβα καλά. Αύριο το πρωί θα μας τα πείτε, το μεσημέρι, πότε. Πριν αύριο το πρωί. Πριν από αύριο. Θα ήταν καλό να τα έχουμε τα κείμενα αυτά πριν ε, τις 9 που θα συναντηθούμε το πρωί αύριο για να προετοιμαστούμε. Well, we, we haven't, we haven't discussed... Δεν το έχουμε συζητήσει, αλλά αν δεν έχουμε τις συμβασικές τροπολογίες, δεν θα έχει νόημα και η συνεδρία των συντονιστών, ε, των σκιωδών, συγγνώμη. Άρα πριν από αύριο, το θα τα έχετε πάρει. Ευχαριστώ, Μπάρτ. Αν ήταν εδώ θα συμφωνούσε ο κύριος Γκίγκολ. Τι είμαι εσύ να ευχαριστήσω τους δύο συνεισηγητές, πολύ δύσκολο θέμα, να ευχαριστήσω και τους άλλους συναδέλφους. Λίγη συνεδρίαση. Ευχαριστώ. Γεια σας.